Eh, Μπορούμε να ξεκινήσουμε με τις εργασίες μας. Η κυρία Μάλστρομ ε, βρίσκεται κάθοδον, αλλά θα ήθελα καταρχήν να κάνω ορισμένες ε, ανακοινώσεις. Όπως ε, γνωρίζετε, βιντεοσκοπείται η συνεδρίασή μας, γι' αυτό θα ήταν σκόπιμο ε, όλοι να καθόσαστε στη θέση σας έτσι ώστε να μπορεί να σας κεντράρει σωστά η τηλεόραση. Χτες στους συντονιστές προβήκαμε στις εξής συστάσεις έτσι ώστε να τις εγκρίνετε. Πρώτον, προετοιμασία των ακροάσεων του, επιτρόπου, του υποψήφιου επιτρόπου ο οποίος θα έχει το χαρτοφυλάκιο Αύκο, έχουμε, θα έχουμε έναν εισηγητή από το ΕΛΚ, τον οποίο θα ορίσουμε. Ε, οριζόντια σύσταση όλων των διαδικασιών, σε αυτή την περίπτωση, η εισηγητής είναι ο συνάδελφος Νταφ. Αυτό μας όρισαν οι πολιτικές ομάδες. Επίσης, εξηγήσαμε, επεξηγήσαμε τη θέση μας σε σχέση με το πρόγραμμα της Στοχόλμης και εγώ θα ασχοληθώ άμεσα με το ζήτημα. Στη συνέχεια προβλέπεται η επίσκεψη μιας, μετάβαση μιας αντιπροσωπείας στη Μαδρίτη στις 2 και 3 Δεκεμβρίου, καθότι έχουμε την Ισπανική Προεδρία το επόμενο εξάμεινο. Θα έχουμε τις ε, πρώτες επαφές, θα έχουμε δύο μέλη από το ΕΛΚ, δύο από τους σοσιαλιστές, έναν από τους φιλελεύθερους και έναν από τους πρασίνους θα ορίσουν, θα προσδιορίσουν τα ονόματα οι ομάδες εν ευθέτω χρόνο. Είχαμε μία μακρά συζήτηση χθες στην Επιτροπή σχολιάζοντας την απόφαση του ε, Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου της Κάρλς Ρούης. Δεν θα ε, οργανώσουμε μια ακρόαση άμεσα, θα προβούμε στις, ανάλογες, στις σχετικές συστάσεις και σχόλια πριν και η νομική υπηρεσία μας παρουσίασε τη θέση της προφορικά στα γερμανικά, άρα η γραμματεία μας θα διευθετήσει το θέμα της μετάφρασης και θα διανεμηθεί σε όλους τους ενδιαφερόμενους. Εάν συμφωνείτε, λοιπόν, μπορούμε να εγκρίνουμε. Εγκρίνουμε την ε, έκθεση των συντονιστών. Νομίζω ότι ο συνάδελφος Μπαρνιέ ζήτησε το λόγο επί του θέματος ή κάνω λάθος. Έχετε το λόγο. Κύριος Μπαρνιέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε επειδή έχουμε αρκετό χρόνο ακόμη μπροστά μας, θέλω να περάσω σε ένα θέμα το οποίο αναφέρατε και αφορά την συζήτηση, την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση που κάναμε χθε για τα σχόλια ή την ανάλυση ή τα πορίσματα από την υπόφαση του δικαστηρίου της Καλσούης. Δεδομένου ότι πρόκειται για ένα πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα και υπάρχουν πολλές αντιπαραθέσεις μεταξύ των ε, εθνικών, τοπικών, ευρωπαϊκών αρμοδιοτήτων τα χαρακτηριστικά με τα κάθε χώρα σε σχέση με την Ευρώπη, πρέπει να πω ότι τα επόμενα πέντε χρόνια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να διαδραματίσει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο για να αποκαταλάβει τις που θα γίνουν, τις πολύ σημαντικές για αυτό το τόσο ουσιαστική σημασία θέμα για όλους. Διαρωτώ με λοιπόν αν εκτός των ε, συνήθων τόπων στο οποίο συζητούμε αυτό το θέμα δεν θα έπρεπε με δική μας πρωτοβουλία το θέμα αυτό να συζητηθεί και σε επίπεδο εθνικών κοινοβουλίων στα πλαίσια της δικής τους Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να προετοιμάσουμε αυτή τη συζήτηση και να δείξουμε ότι ε, δεν μας ενοχλεί το θέμα αυτό και η δυσκολία που ενέχει. Θα πρέπει λοιπόν να οργανωθούμε τα επόμενα πέντε χρόνια στις 27 πρωτεύουσές μας, ώστε να συζητηθεί αυτό το θέμα, λαμβάνοντας υπόψη την κατανομή των αρμοδιοτήτων στα πλαίσια της συνθήκης Λισαβόνας. Το λέγω αυτό, είναι μια υπόδειξη, μια πρόταση και δεν ήθελα να το σκεφτούν οι συντονιστές. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για αυτή την υπόδειξη. Πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η υπόδειξη, κρίνω, διότι η χτεσινή συζήτηση αφορά την ταυτότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε ενώπιόν μας ε, μια εργασία η οποία είναι χρονοβόρα Ε, δεν θα προβούμε σε, στην επίκριση της απόφασης του Συνταγματικού Δικαστηρίου, αλλά θα πρέπει να προβούμε σε μια γενικότερη σκέψη. Μπορούμε να μεταβούμε σε όλες τις πρωτεύουσε και έχοντας μπροστά μας πέντε χρόνια έχουμε πολλή δουλειά. Έφτασε η υπουργό. Δεν θα ήθελα να ανοίξουμε τη συζήτηση τώρα όμως. Θεωρώ ότι αυτή η συζήτηση είναι άκρος ενδιαφέρουσα. Α, έφτασε η αναπληρώτρια υπουργός. Ringraziamo. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Υπουργό Τσιτσίλια Μάλστρομ. Δεν ξέρω κατά πόσο προφέρω σωστά το όνομά σας. Την κυρία Μάλστρομ, λοιπόν, την οποία γνωρίζετε πολύ από εσά, διότι ήταν συνάδελφος στο παρελθόν. Ήδη την γνωρίζετε πολύ από εσά διότι ήταν ευρωβουλευτής από το 1999 στο 2006 και μία αντιπροσωπεία μας μετέβη στη Στοκχόλμη και ήρθε σε είχε επαφές και με τον Πρωθυπουργό. Εσείς ήσασταν επικεφαλής και μεταβήκατε και αρκετοί από εσά. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα που βρίσκεστε εδώ Ελπίζουμε να έχουμε και άλλες ευκαιρίες να συναντηθούμε πριν από το τέλος της Προεδρίας σας, εδώ στις Βρυξέλλες. Και χαιρόμαστε ιδιαίτερα γιατί μπορούμε να σας ακούσουμε για το πρόγραμμα της Σουηδικής Προεδρίας, γιατί μας απασχολεί ιδιαίτερα, με βάση τις αρμοδιότητες αυτής της Επιτροπής, μας απασχολεί ε, ιδιαίτερα το δημοψήφισμα στην Ιρλανδία και αν η συνθήκη της Λισαβόνας κυρωθεί, θα θέλαμε να καταρτήσουμε τις σωστές κατευθυντήρες γραμμές για να τεθεί σε εφαρμογή. Βεβαίως, υπάρχει και το σοβαρό πρόβλημα του διορισμού του Πρόεδρου της Επιτροπής. Είναι ένα θέμα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε σύντομα και ελπίζουμε ότι η Σουηδική Προεδρία θα μας βοηθήσει και επ' αυτού. Όχι μόνο στον ορισμό του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά στη σύνθεσή της γενικότερα. Θα θέλαμε λοιπόν να εκφράσετε τις απόψεις σας και στη συνέχεια θα ανοίξει η συζήτηση με ερωτήσεις και απαντήσεις. Σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά κυρία Μάλστρομ και έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, herr eh, Πρόεδρε, κύριοι βουλευτές, είναι ιδιαίτερη τιμή για εμένα να βρίσκομαι εδώ καθώς ήμουν και στο παρελθόν Ευρωβουλευτής και μάλιστα μέλος αυτής της ε, Επιτροπής για αρκετές ε, θητείες. Οπότε θα ήθελα πρώτα απ' όλα να συγχαρώ τον κύριο Κασίνη για την ε, Προεδρία του και θα ήθελα να συγχαρώ και όλα τα μέλη της Επιτροπής για την εκλογή τους. Ξέρετε πως έχουμε ακόμη τέσσερις μήνες που απομείνει στην Σουηδική Προεδρία και αναμένουμε με αγωνία την συνέχεια. Αυτό το οποίο είδαμε στις ευρωεκλογέ είναι ένα ορόσημο της ευρωπαϊκής ε, συνεργασίας. 20 χρόνια μετά το 1989 πολίτες ε, των 27 κρατών μελών ψήφισαν ταυτόχρονα. Ποιος θα μπορούσε να είχε φανταστεί κάτι τέτοιο για τους πολίτες όλων αυτών των χωρών να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα και να ψηφίσουν ελεύθερα τους εκπροσώπους τους σε ένα δημοκρατικό κοινοβούλιο. Μάλιστα, εάν ε, ανατρέξουμε στην ε, ιστορία, θα δούμε πως ε, σήμερα η σήμερα, σαν σήμερα ξεκίνησε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, υπάρχουν και εκδηλώσεις σχετικές στην Πολωνία. Στην χώρα μου υπήρχε αρκετά μεγάλη συμμετοχή στις ευρωεκλογέ άνω του 45%. Δυστυχώς πανευρωπαϊκά υπήρχε μείωση του ποσοστού συμμετοχής στις εκλογές, οπότε θα πρέπει να αναρωτηθούμε γιατί οι πολίτες μας απέχουν από τις ε, ευρωεκλογές για να αναδείξουν το εξαίρετο αυτό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βεβαίως ε, αντιλαμβάνομαι πως ε, υπάρχει τώρα αναθεώρηση των διατάξεων που αφορούν την εκλογή των μελών που Βεβαίως ε, έχουν μείνει αναλύτως από το 1976 και μάλιστα είναι κάτι που έχει αναλάβει ο Άντριου Νταφ. Η Σουηδική Προεδρία επίσης έχει αναλάβει μια σχετική πρωτοβουλία. Οι πολίτες μας περιμένουν πολλά από εμά. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει με την πιστοτική κρίση, με την αυξανόμενη ανεργία που πλήττει όλα τα κράτη-μέλη. Επίσης θα πρέπει να ανταποκριθούμε στην πρόκληση της κλιματικής αλλαγής. Οπότε όλα αυτά θα κυριαρχήσουν στην δουλειά μας καθ' όλη τη διάρκεια του φθινοπόρου και είναι πολύ φιλόδοξο το να θέλουμε να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα ζητήματα. Πρέπει να ενισχύσουμε και την ανταγωνιστικότητά μας για να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας και να έχουμε μια υφόρα ανάπτυξη και καλύτερο περιβάλλον. Τώρα, θα πρέπει να εγκρίνετε εσείς και τον νέο πρόεδρο της Επιτροπής και μια ολόκληρη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προφανώς δεν ξέρουμε τι γίνεται ακόμα με την συνθήκη της Λισαβόνας. Θα τεθεί ενισχύ επί Σουηδικής Προεδρίας. Εάν γίνει όντως δεν έχουμε πολύ καιρό στη διάθεσή μας για να γίνουν αυτές οι θεσμικές αλλαγές οι οποίες χρειάζονται. Θα πρέπει εμείς να προσπαθήσουμε να διευκολύνουμε τη μετάβαση από την παλαιά στην νέα συνθήκη. Οπότε, όπως σας είπα, θα βασιζόμαστε στον διάλογο και τη στενή συνεργασία μαζί σας, γιατί πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία όσο περισσότερο γίνεται. Το πρόγραμμα της Προεδρίας μας αποτελεί μέρος ενός προγράμματος 18 μηνών που είχαμε συμφωνήσει και με τους Γάλλους εναδέλφους από την προηγούμενη Προεδρία και θέλουμε πράγματι να διαφυλάξουμε τα συμφέροντα της Ένωσης συνολικά και των πολιτών μας. Θέλουμε να αποκαταστήσουμε επίσης την εμπιστοσύνη στις χρηματαγορές, να υπάρχει μια επίβλεψη των αγορών η οποία θα λειτουργεί, να δούμε κάποιες μακροπρόθεσμες λύσεις για βιώσιμη ανάπτυξη που θα εγγυάται απασχόληση και ευημερία ακόμα και ε, κατά την εποχή αυτή του αυξημένου παγκόσμιου ανταγωνισμού. Και αυτό θα έλεγα πως χαρακτηρίζει όλες τι δραστηριότητε μα σε όλους τους συνδυασμού του Συμβουλίου. Θέλουμε να ξαναδούμε τη στρατηγική της Λισαβόνας και πράγματι γεγονό είναι πως αυτέ οι συζητήσει θα ολοκληρωθούν επί Ισπανικής Προεδρίας. Η κλιματική αλλαγή είναι μια μεγάλη πρόκληση που αντιμετωπίζουμε. Δεν έχουμε χρόνο να χάσουμε, αλλά δεν μπορούμε να επιτύχουμε και μόνοι μας ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να καταλήξουμε σε κάποια θετικά επιτυχή βήματα στην Κοπενχάγη μετά τις θετικές εξελίξεις τους ε, G8 για πρώτη φορά είχαμε μια αποδοχή για να έχουμε μια οροφή αύξησης της θερμοκρασίας 2 βαθμών Κελσίου. Όπως σας είπα πρέπει να δούμε πώς θα καταλήξουμε σε μια πιο ασφαλή και πιο ανοιχτή Ευρώπη. Έχουμε επίσης ένα πενταετές πρόγραμμα ε, συνεργασία το λεγόμενο πρόγραμμα της Στοκχόλμης καθώς και μια στρατηγική για την βαλτική και την περιφερειακή συνεργασία που ελπίζουμε ότι θα αποτελέσει υπόδειγμα και για άλλες περιοχές. Επίσης σκοπεύουμε να θέσουμε τις ε, βάσεις για την ειρήνη, τη δημοκρατία και του σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανά την Ιφίλιο για να διασφαλίσουμε βέβαια και την ευημερία και την ειρήνη στην Ευρώπη και στο μέλλον. Ένα από τα ερωτήματα τα οποία μας απασχολεί είναι το τι πρέπει να κάνουμε ως Προεδρία. Ελπίζω να έχετε την ευκαιρία να επισκεφτείτε την ε, σελίδα μας. Ελπίζω να είναι ως το δυνατόν πιο προσβάσιμη στους ε, πολίτες, κάτι το οποίο μας απασχολεί ιδιαίτερα με βάση την μειωμένη συμμετοχή σε ευρωεκλογέ. Ε, επίσης πρέπει να δούμε και τους κανόνες για την δημοσίευση των εγγράφων, την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα. Ξέρω πως η Επιτροπή Ελευθεριών θα παίξει τον βασικό ρόλο εδώ πέρα, αλλά γνωρίζω πως και η ειδική επιτροπή θα το παρακολουθήσει στενά το θέμα. Τον Ιούνιο επιτύχαμε μια συμφωνία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την νομική εγγύηση που δόθηκε στην Ιρλανδία αλλά και για να οριστεί εκ νέου ο κ. Μπαρόσο, πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επιπλέον ε, θα πρέπει να τεθεί ενισχύ η συνθήκη της Λισαβόνας πριν από το τέλος του έτους. Η απόφαση τώρα για τις εγγυήσει που δόθηκαν στην Ιρλανδία στόχο είχε να ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Πρέπει να δούμε επίσης ε, το τι γίνεται με την φορολογία και την Ιρλανδική ουδετερότητα και ελπίζουμε έτσι να καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε την σύμφωνη γνώμη της Ιρλανδίας για την συνθήκη της Λισαβόνας. Νομίζω πως ε, έχει κάνει πολύ καλή δουλειά η Ιρλανδική κυβέρνηση. Η απόφαση αυτή είναι νομικά δεσμευτική και θα τεθεί ενισχύ ταυτόχρονα με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Στην ε, συνεδρίαση του Ιουνίου το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε πως τον Δεκέμβριο, υπό την προϋπόθεση πως θα είναι ενισχύ η συνθήκη της Λισαβόνας, να ληφθεί μια απόφαση έτσι ώστε η Κομισιόν να συνεχίσει να έχει ένα μέλος από κάθε κράτος μέλος γιατί αυτό ήταν σημαντικό για την Ιρλανδία γιατί όπως ξέρετε μέχρι στιγμής έχει εγκριθεί σε 23 κράτη-μέλη η συνθήκη έχει επικυρωθεί στην Πολωνία, Τσεχία και Γερμανία έχει προχωρήσει η επικύρωση αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί ολόκληρη η διαδικασία οπότε γνωρίζουμε πως έχουμε ακόμα και ένα δημοψήφισμα στην Ιρλανδία τον Οκτώβριο. Ελπίζω πραγματικά το αποτέλεσμα να είναι θετικό για τη συνθήκη της Λισαβόνας, γιατί έτσι θα γίνει πιο ανοιχτή, αποτελεσματική και δημοκρατική η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα μας δώσει μεγαλύτερη επιρροή στην ε, διεθνή σκηνή. Τώρα, η συναπόφαση είναι πάρα πολύ σημαντική στο νομοθετικό πλαίσιο θα αυξηθούν οι αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου, θα ευαθυνθεί έτσι η δημοκρατία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη του κόσμου προς την Ένωση. Τώρα παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον την συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την συνθήκη τη Λισαβόνα. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Γιολάνη, τον τον Έλα και λοιπού για το έργο τους. Είμαι διατεθειμένη να ξεκινήσω το προπαρασκευαστικό έργο για να έχουμε μια νέα συνθήκη. Ξέρω πως πρέπει να ληφθούν πάρα πολλές αποφάσεις τη μέρα την οποία θα τεθεί ενισχύ η συνθήκη. Πρέπει να έχουμε προετοιμαστεί από πριν. Αυτό σημαίνει πως Συμβούλιο και Κοινοβούλιο θα πρέπει να συμφωνήσουν σε κάποια πράγματα. Παραδείγματος χάρη το πως θα αντιμετωπίσουμε τις νομοθετικές προτάσεις ε, στους τομείς εκείνους στους οποίους θα έχουμε συναπόφαση αλλά δεν έχουμε ακόμα αυτή τη στιγμή. Επίσης κάτι άλλο που θα είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν τεθεί ενισχύ η συνθήκη. 80 α, βουλευτές θα έχουμε από κράτη τα οποία θα γίνουν ε, κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε ελπίζω να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα ζήματα, να μπορέσουμε να έχουμε κάποια μεταβατικά μέτρα μέχρι να τεθεί ενισχύ η συνθήκη το 2010. Επίσης, εξετάζουμε το ζήτημα ακριβώς αυτό του τι θα γίνει με τους ε, παρατηρητές αυτή τη στιγμή ε, τεθεί ενισχύ η συνθήκη και πριν ληφθεί η απόφαση για τους μεταβατικούς κανόνες. Επίσης η κοινή ε, εξωτερική υπηρεσία που θα είναι ένας ρόλος θα μοιράζονται κομισιόν και συμβούλιο για να εκπροσωπήσουν την Ένωση σε παγκόσμιο επίπεδο. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει σε επίπεδο εμπορίου, διεύρυνσης, ανάπτυξης κλπ πρέπει τα ζητήματα αυτά να μας απασχολούν διαρκώς γιατί αυτά καθορίζουν τη σχέση μας με τον υπόλοιπο κόσμο. Η απόφαση για την υπηρεσία εξωτερικής δράσης είναι κάτι που επεξεργαζόμαστε αυτή τη στιγμή πρέπει να γίνει πραγματικότητα το συντομότερο δυνατόν μόλις τεθεί η συνθήκη της Λισαβόνας και πρέπει να δούμε και τον ρόλο του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αυτός ή αυτή θα είναι υπεύθυνο για την διαχείριση της ημερήσιας διάταξης του Συμβουλίου, την εφαρμογή της και την εκπροσώπηση της Ένωσης στον έξω κόσμο. Οπότε επανερχόμαστε τώρα στο τι θα γίνει εάν δεν τεθεί ενισχύ τη συνθήκη της Λισαβόνας ή εάν έχουμε και άλλες καθυστερήσεις. Προφανώς δεν θέλουμε να συμβεί αυτό, αλλά ε, παρόλα αυτά η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να λειτουργεί με βάση τη συνθήκη τη νίκη. Προφανώ εμεί θέλουμε μια πιο ανοιχτή και αποτελεσματική Ευρώπη, αλλά θα πρέπει να εργαστούμε με βάση τη συνθήκη, την εκάστοτε συνθήκη που ισχύει. Θα πρέπει να οριστεί λοιπόν μια νέα επιτροπή και να δούμε το τι μπορούμε να κάνουμε με την συνθήκη που ισχύει αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίσουμε όπως είπα το οργανωμένο έγκλημα, την κλιματική αλλαγή κτλ. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να ξεκινήσει τα καθηκοντά της, να αναλάβει τα καθηκοντά της πάρα πολύ γρήγορα η νέα Κομισιόν για να μην κολλήσουν τα πράγματα. Δεν μπορούμε αλλιώς να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στην Ευρώπη. Ελπίζω πως στην Ολομέλεια του Σεπτεμβρίου το Κοινοβούλιο θα αποφασίσει να συμφωνήσει στον ε, οριστεί ο κύριος Μπαρός ως πρόεδρος της Επιτροπής και μετά θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στον διορισμό της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εάν λοιπόν τεθεί η συνθήκη της Λισαβόνας θα έχουμε ένα επίτροπο ανακράτος μέλος, εάν είναι η συνθήκη της Νίκης θα έχουμε λιγότερους επιτρόπους. Θα πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε. Τα πάντα εξαρτώνται από το δημοψήφισμα της Ιρλανδίας. Μόλις ε, λάβει απόφαση βεβαίω το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τον αριθμό των μελών θα υποβάλουμε την απόφασή μας αμέσως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να μπορέσετε να κάνετε και εσείς τις ακροάσεις το συντομότερο δυνατόν. Η Επιτροπή θα πρέπει να δει μια σειρά προκλήσεων, να δούμε το θέμα της 1ης ε, Νοεμβρίου. Πράγματι θα πρέπει να υπάρχει μια υπηρεσιακή κομισιόν τρόπον τι να. Ε, προφανώς η κατάσταση είναι εξαιρετική, αλλά όλοι έχουμε συμβόλαιο και έχουμε ευθύνη, με συμβούλιο και κοινοβούλιο να φροντίσουμε να κυλήσουν τα πράγματα όμαλα. Επίσης θα υπάρξει και ύπατος εκπρόσωπος για την ΚΕΠΑ εντεθεί, ε, όπως είπα, ενισχύει η συνθήκη και θα υπάρχει και αρμόδιος για τις εξωτερικές σχέσεις. Οπότε και εδώ πέρα έχει σημαντικό ρόλο να παίξει το Κοινοβούλιο. Πριν οριστεί αυτός ο ύπατος εκπρόσωπος, οπωσδήποτε η Προεδρία θα έρθει σε επαφή με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αυτό σημαίνει πως ο ύπατος αυτός εκπρόσωπος ε, θα μπορέσει να αναλάβει ε, τα καθήκοντά του αμέσως μόλις τεθεί εν ισχύ η συνθήκη. Επίσης 10 Οκτωβρίου θα έχουμε συμβόλαια και συμβούλια με και 11 και 12 Δεκεμβρίου οπότε θα συζητήσουμε τον Οκτώβριο τους ε, διορισμούς, όπως όπω είπα, των μελών της ε, Κομισιόν, αλλά προφανώς θα πρέπει να γίνει και μια συζήτηση για διάφορα θεσμικά θέματα και στην ε, Σύνοδο Κορυφής του Δεκεμβρίου. Οπότε το πρόγραμμα μας είναι γεμάτο, ελπίζουμε πως η νέα συνθήκη θα τεθεί ενισχύ προσεχώς για να γίνει πιο προσβάσιμη στους πολίτες της Ευρωπαϊκή Ένωση και χρειάζεται σκληρή δουλειά για να προετοιμάσουμε την κατάσταση. Πρέπει όλοι μας λοιπόν να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και τα τρία θεσμικά όργανα και αντιλαμβάνομαι πως είστε έτοιμοι να αναλάβετε αυτές τις ευθύνες και εγώ θέλω να συνεργαστώ στενά με την Επιτροπή σας και το Κοινοβούλιο για το υπόλοιπο της Προεδρίας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μου δώσετε την ευκαιρία να μιλήσω εδώ σήμερα και είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Σας ευχαριστούμε, κυρία Υπουργέ. Ακούσαμε μία πλήρη, έναν πλήρη απογραφικό κατάλογο των ε, ευθυνών και των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συνθήκη της Λισαβόνας, εάν τεθεί σε ισχύ. Έχουμε πολύ μεγάλη εργασία μπροστά μας και αυτό αφορά τη δική σας Προεδρία, τις επερχόμενες, αλλά και τη δική μας Επιτροπή. Θα λάβουμε υπόψη πολύ σοβαρά τις υποδείξεις σας για την επίλυση προβλημάτων που προβλέπουν, προβλημάτων προβλέπονται και από τη συνθήκη της Λισαβόνας. Θα ήθελα τώρα να παρέμβουν οι συνάδελφοι. Ήγο, Fox και ε, Δίνω το λόγο λοιπόν στον Μέντες Δεβίγκο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλώς ορίσατε. Και πάλι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ξέρω ότι μιλάτε τέλεια και τη γλώσσα μου. Ξέρω με τους ομάδες μου θα σας πω ότι χαίρομαστε που είστε και πάλι εδώ. Ξέρω ότι ήταν μεγάλη απώλεια για μας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να φύγετε, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή τη ε, στιγμή έχετε ένα εξαιρετικό ρόλο ασκώντας στην Προεδρία. Θέλω να σας κάνω την εξή ερώτηση. Σήμερα το πρωί μπήκα στην ιστοσελίδα σας και βρήκα πολλές απαντήσεις στα θέματα τα συνταγματικά που μας απασχολούν. Γι' αυτό θα περιοριστώ μόνο σε ένα σχόλιο και σε μία ερώτηση. Και έτσι θα έχουμε περισσότερο χρόνο οι συνάδελφοι για να σας κάνω ερωτήσεις. Το σχόλιο είναι το εξή. Εάν υπάρχει κάποιο άτομο το οποίο έχει να διαδραματίσει ρόλο πάρα πολύ ευαίσθητο στα πλαίσια της ε, συλλογικού οργάνου που είναι η Επιτροπή, είναι ο ύποπτος εκπρόσωπος. Η πρόταση λοιπόν αυτή έχει γίνει και ξέρω ότι υπάρχει, πρέπει να υπάρχει για την ε, τελική ψηφοφορία του συνόλου των επιτρόπων πάρα πολύ καλή επικοινωνία για να ξέρουμε ποιο θα είναι η προσωπικότητα που θα ασκήσει αυτό το, ε, θα οριστεί ως ε, εκπρόσωπος και θα μας βοηθήσει η καλή επικοινωνία να βρούμε απαντήσεις στις ερωτήσεις μας. Η ερώτησή μου αυτή είναι το αυτό το σχολείο. ερώτηση. Τι γίνεται με τις ε, εξωτερικές υπηρεσίες της Κομισιόν. Πού βρισκόμαστε. Το θέμα αυτό είναι ένα θέμα ουσιαστικής σημασίας και ξέρω ότι δεν θα ασχοληθείτε εσείς εξ ολοκλήρου, θα περάσει και στη δική μας την αρμαδιότητα στην επόμενη Προεδρία. Πού βρισκόμαστε λοιπόν με το θέμα αυτό του του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ Σεσίλια. Κύριος ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Μάλστρομ για την παρέμβασή σας, για την παρουσία σας και για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Σημερίζομαι το κύριο πνεύμα και τις ιδέες που εκφράσατε στις παρεμβάσεις και εξονόματος της σοσιαλιστικής ομάδας. Θα ήθελα να πω ότι έχουμε κάποια ερωτηματικά και κάποιες ανησυχίες τις οποίες θα ήθελα να εκφράσω. Πρώτα απ' όλα, κάτι που έχει σχέση με την δικές σας αρμοδιότητες. Τι θέλετε κατά βάθος. Να τεθεί σε εφαρμογή η συνθήκη της ε, Λισαβόνας και να δει μια ε, ουσιαστική όθη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά την άποψή σας, όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία υποψηφίσματος στην Ιρλανδία, δεν θα υπάρχει άλλο πρόβλημα. Έχετε κάποιες επαφές με την τσεχική Προεδρία. Διότι όταν θα ξεπεράσουμε αυτό το μεγάλο εμπόδιο που θα είναι το δημοψήφισμα στην Ιρλανδία, δεν θα έχουμε άλλο. Τι κάνετε εσείς για να εξασφαλίσετε ότι δεν θα υπάρχουν μεγάλα προβλήματα εκ των Δεύτερη ερώτηση, που έχει σχέση με κάτι το οποίο επίσης θεωρώ σημαντικό. Άκουσα και διάβασα τις δηλώσεις που κάνετε σε σχέση με την σημασία που έχει για την Ευρωπαϊκή Ένωση η επικύρωση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο της πρότασης την οποία υπέβαλε το Συμβουλίο. Βεβαίως, 27 χώρες να αποφασίσουν με ομοφωνία ε, στα πλαίσια του Συμβουλίου του Ιουνίου και να μας βάλουν πρόβληση ήταν σημαντικό. Έχουμε όμως κάποιες αμφιβολίες και σε όλες τις ομάδες εκτός από το ΕΛΚ υπάρχουν μεγάλες ε, αντιφάσεις για τον τρόπο με τον οποίο και ερωτηματικά για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να γίνει αυτή η επικύρωση. Σας ερωτώ λοιπόν πώς θα μπορούσατε να πείσετε τους ευρωβουλευτές που θεωρούν ότι είναι καλύτερο να κυρωθεί ή ε, όχι ο Μπαρόσο ήδη με, ε, ε, όταν θα έχει κυρωθεί η συνδίκη της ή πριν. Και αυτά στα πλαίσια της δικής σας προεδρίας. Γιατί αυτό είναι ένα θέμα το οποίο άπτεται όλων των συζητήσεων που κάνουν. Υπάρχουν κάποιοι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που απαιτούν κύρωση ή όχι του Προέδρου της Επιτροπής και του συνόλου των Επιτροπών να γίνει όταν θα έχει τεθεί σε εκκίνηση η συνθήκη της Λισαβόνας. Το Συμβούλιο μας είπε αρχίστε από τώρα αυτή τη διαδικασία. Ήδη θέλανε να γίνει κάτι τέτοιο τον Ιούλιο. Αρνήθηκε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είπαμε ίσως το Σεπτέμβριο. Αλλά η διάσκεψη των Προέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να πάρει κάποια απόφαση στις 10 Σεπτεμβρίου εάν ναι ή όχι κάτι τέτοιο θα γίνει στη Σύνοδο Σεπτεμβρίου. Η ερώτησή μου λοιπόν κυρία Μάλστρομ είναι για το Συμβούλιο σε ποιο μέτρο είναι σημαντικό να γίνει αυτή η κύρωση από το Κοινοβούλιο και γιατί δεν θα πρέπει να περιμένουμε τη, να ισχύσουν οι κανόνες εφαρμογής συνθήκης της Λισαβόνας. Μια τρίτη ερώτηση. Η αναφορά στην θεσμική ισορροπία μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Επιτροπής. Ξέρετε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκφράστηκε υπέρ του συσσωροπίας στην εξωτερική αυτή υπηρεσία όπως λέγεται. Έτσι όπως λέγεται αυτή η εξωτερική υπηρεσία ελέγχθη ότι θα πρέπει, και αυτό είναι κάτι το οποίο είπαμε και εμείς, να είναι μέρος της Επιτροπής. Ποια είναι όμως η άποψη του Συμβουλίου για αυτό το θέμα και πώς θα μπορέσει να γίνει σεβαστή η συνταγματική η θεσμική ισορροπία. Κάτι άλλο το οποίο μας απασχολεί όλους επίσης. Σε κάποιες χώρες, και στη χώρα σας και στη δική μου, η συμμετοχή στις ευρωπαϊκές εκλογές μετρίως καλή ήταν. Σε άλλες χώρες ήταν καλύτερη, όπως το Βέλγιο. Αλλά συνειδητοποιούμε ότι υπάρχει μια επικίνδυνη τάση να μην ενδιαφέρονται οι Ευρωπαίοι πολίτες για το τι ακριβώς γίνεται εδώ και να αδιαφορούν για τις ευρωεκλογέ. Και κάθε Όλο και περισσότερο υπάρχουν ευρωσκεπτικιστέ ή αντιευρωπαίοι, αντι... ενάντι στην ευρωπαϊκή ιδέα. Όλο και περισσότερο το συνειδητοποιούμε αυτό. Εκτός λοιπόν από αυτό που προκαλεί ανησυχία, υπάρχουν στο Συμβούλιο προτάσεις ή πρωτοβουλίες για να μπορέσουμε κατά κάποιο τρόπο να λύσουμε αυτό το δομικό πρόβλημα που έχουμε, το διαρθρωτικό πρόβλημα που έχουμε με την ε, Ευρώπη. Η ιδέα της ΕΕ ενθουσίασε πάρα πολλά εκατομμύρια πολιτών εδώ και χρόνια, αλλά αυτή τη στιγμή αλλά έχουν αλλάξει τα πράγματα. Κάτι άλλο να ερωτήσω επίσης. Στο Βούλιο, στα πλαίσια της στρατηγικής έχετε ποτέ σκεφτεί την ε, ανανέωση όλες τις διαδικασίες Λισαβόνες. Πρόκειται για ένα εξαιρετικό όνειρο. Το 2000 οι Ευρωπαίοι θέλησαν να γίνει η Ευρώπη το πιο ανταγωνιστικό μέρος του κόσμου με εξαιρετική ποιότητα, με τρομερή κοινωνική συνοχή, με τις καλύτερες συνθήκες εργασίας κτλ. Όνειρο ήτανε όμως, γιατί δεν είδαμε τα τελευταία δέκα χρόνια να ολοκληρώνουν τα πράγματα. Δεν προχωρήσαμε. Σχεδόν καθόλου. Το ερώτημα μου είναι, μετά από δέκα χρόνια, αφού είδαμε ότι δεν ολοκληρώθηκαν οι στόχοι, δεδομένου ότι αύριο έχουμε 2010, στα πλαίσια της Προεδρίας, στο Συμβούλιο γίνεται κάποια συζήτηση για την ανανέωση της στρατηγικής Λισαβόνας. Και τελειώνω τώρα και συγγνώμη που μακρηγόρησα. Το επόμενο ερώτημά μου είναι το εξή. Τα μέσα που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι επαρκή ή όχι. Είπατε εσείς ότι ο μεγάλος αντικειμενικός στόχος της Σουηδικής Προεδρίας όπως και άλλων προεδριών είναι να βγάλουμε την Ευρώπη από την ε, κρίση. Έχει καλώς. Σωστό αυτό, αλλά έχουμε τα κατάλληλα μέσα. Πραγματικά η Ευρώπη κάνει τίποτα περισσότερο από το να μας συντονίζει με, με γλέτες τις οποίες ε, κάνει. Έχουμε τα επαρκή οικονομικά και νομισματικά μέτρα. Ε, έχετε την εντύπωση, η Προεδρία η Σουηδική, το Συμβούλιο, έχετε όντως την εντύπωση ότι έχουμε ένα επαρκές οικονομικό και εκτελεστικό μέσων το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε για να βγούμε από την κρίση. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ντάφ έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχήν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Σεσίλια και να τη συγχαρώ. Υποθέτω ότι απολαμβάνει την Προεδρία Σεσίλια Δεν μας το είπες αυτό. Ίσως μας το πεις όταν απαντήσεις στις ερωτήσεις. Ως προς το θέμα του διορισμού του Προέδρου της Επιτροπής, ο κύριος Καοριγκή ανέφερε ότι η διαδικασία ε, είναι ιδιαίτερα ταχεία. Δεν μπορεί να κατηγορηθεί το Κοινοβούλιο ότι προσεγγίζει αυτό το θέμα με σπουδή. Νομίζω ότι ήταν πολύ σωστό το ότι αναβάλαμε την απόφαση από τον Ιούλιο στο Σεπτέμβριο, για το Σεπτέμβριο, έτσι ώστε όλοι μας να πάρουμε μία βαθιά ανάσα και να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα πιο σοβαρά από ότι τον Ιούλιο. Τα θέματα δηλαδή που θα απασχολήσουν, ως προς τα θέματα που θα απασχολήσουν την Προεδρία της Επιτροπής. Με εξέπληξε το γεγονός ότι η δυνάμη της συνθήκης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να συνεργαστεί με το Συμβούλιο έτσι ώστε ο διορισμός της Επιτροπής να διενεργηθεί αποτελεσματικά. Και είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι ότι ακολουθούμε τη σωστή οδό. Θα πρέπει να κινηθούμε δυνάμει των όρων της παρούσα συνθήκης. Της παρούσας συνθήκης. Μέχρι ότου δούμε ε, ποιος δρόμος ε, διανοίγεται με τη νέα συνθήκη που θα τεθεί σε ισχύ. Νομίζω ότι θα ήταν ε, απαράδεκτη η κολλησιεργία και βέβαια θα παραβαίναμε και τη συνθήκη αν γινόταν διαφορετικά. Ελπίζω λοιπόν να μπορέσουμε να κινηθούμε ε, τάχιστα το Σεπτέμβριο και να εγκρίνουμε τον διορισμό του Πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε σχέση με τον διορισμό του Πρόεδρου του Συμβουλίου, θα ήθελα να ρωτήσω το εξής. Πιστεύετε ότι είναι δυνατός ο διορισμός κατά, την, κατά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου. Δεν αναζητώ ονόματα αυτή τη στιγμή, αλλά θα μας ενδιέφερε να μάθουμε ποιες ε, είναι οι προθέσεις της Σουηδικής Προεδρίας για τον διορισμό του Πρόεδρου του Συμβουλίου. Προτιμάτε κάποιον άνθρωπο τύπου Σαρκοζή ή κάποιον ε, πιο μετριόφρονα πρόεδρο. όπως ισχύει στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να εκφραστεί ως προς την μορφή του Προέδρου του Συμβουλίου. Δηλαδή, τι είδους πολιτικό πρόσωπο προτιμάμε. Αν και η επιλογή είναι προνόμιο του ιδίου του Συμβουλίου. Τρίτον, κατά τη διενέργεια του δημοψηφίσματος στην Ιρλανδία, αν και νομίζω ότι η εκστρατεία αποτελεί βελτίωση, ποιοτική βελτίωση σε σχέση με το προγενέστερο δημοψήφισμα, νομίζω ότι υπάρχουν πολλά ψευδοδιλήμματα που θέτουν οι αντιτιθέμενες δυνάμεις. Δηλαδή το φάσμα του Τούρκου αγρότη, ο οποίος θα οδηγήσει στην κατάρρευση της ΚΑΠ, εάν η συνθήκη της Λισαβόνας τεθεί σε ισχύ. Ποια είναι η προσέγγιση της Σουηδικής Προεδρίας ως προς την ίδια την εκστρατεία. Πιστεύω ότι θα πρέπει να απομακρυνθούμε από αυτό το ψευδοφάσμα του Τούρκου αγρότη. Πολύ ταχύτερα από ό,τι καταφέραμε να απομακρύνουμε το φάντασμα του Πολωνού υδραυλικού κατά την ε, Γαλλική Προεδρία του 2005. Βεβαίως όλοι ελπίζουμε η συνθήκη να τεθεί σε ισχύ. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πολλαπλασιάσουμε την ισχύ της συνθήκης εν μία νυχτή το κοινό μας έχει μετατραπεί σε ένα πολύ ε, κοινικό κοινό σε σχέση με αυτή την κολυσιεργία της ε, κύρωσης της συνθήκης και γι' αυτό θα πρέπει να προωθήσουμε την κύρωση ε, με μία πανηγυρική εκδήλωση έτσι ώστε να δείξουμε ότι η Ευρώπη γυρίζει σελίδα ως προς τις πολιτικές της, την πολιτική της ανέλυξη. Και εάν αναζητάτε τον τόπο Μπορώ να σας προτείνω την Πράγα για να γίνει κάτι τέτοιο. Για να γίνει αυτή η πανηγυρική εκδήλωση. Ευχαριστούμε. Ο συνάδελφος, ο κύριος Φόξ, έχει το λόγο. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ, και σας ευχαριστώ που ήρθατε να μας μιλήσετε σήμερα. Όσον αφορά τον ορισμό του Προέδρου της Επιτροπής η ομάδα μου θεωρεί πως θα πρέπει να προχωρήσετε με την υπόθεση πως ισχύει η συνθήκη της νίκαιας εκτός εάν και μέχρι τη στιγμή που θα επικυρωθεί η συνθήκη της ε, Λισαβόνας και κάποιος συνάδελφος είπε πως ε, ε, ίσως υπάρχει μια αναβλητικότητα που δεν χρειάζεται. Ελπίζω στον ορισμό της Κομισιόν να προχωρήσετε σύμφωνα με την ισχύουσα συνθήκη της νοικίας και εάν ή όταν ισχύσει η συνθήκη της Λισαβόνας τότε θα ληφθούν υπόψη οι διατάξεις της όσον αφορά τον ορισμό του Προέδρου του Συμβουλίου. Η Βαρόνι Κίνοκ, η Βρετανή Υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, κατέστησε σαφέ πω η Βρετανική κυβέρνηση θα υποστηρίξει την υποψηφιότητα του Τόνι Μπλερ. Θα ήθελα να ακούσω τις δικές σας απόψεις ε, και αν θεωρείτε πως τον αποστηριχτή συγκεκριμένο συγκεκριμένος ο βοηθάει την υπόθεση και αν καλωσορίζετε την προοπτική ενός Προέδρου Μπλερ. Εμείς θεωρούσαμε πως ήταν αρκετά αποκρουστικό το να έχουμε Πρωθυπουργό τον Μπλερ, πόσο μάλλον Πρόεδρο του Συμβουλίου. Είναι κάτι που μας γεμίζει τρόμο. Δεν ξέρω αν η εικόνα, το φάσμα, ε, η προοπτική αυτή επηρεάσει τους Ιρλανδούς ψηφοφόρους. Τώρα, για να σοβαρευτώ λίγο για το σχόλιο σας για την ειρήνη, τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα ήθελα να σας ζητήσω να σχολιάσετε σύντομα την κατάσταση στην Γερμανία και το εάν ε, ε, είναι πρόθεσή σας να κάνετε κάτι για την φρικτή κατάσταση εκεί και για το αν μπορούμε να βοηθήσουμε κάποιο τρόπο την Σάνξουτσι και αν αυτό αποτελεί η προτεραιότητα της Προεδρίας. Σας ευχαριστώ. Thank you, President. Ευχαριστώ. And thank you for coming. Ευχαριστώ Κύριε, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Στην αρχική σας παρουσίαση, συγγνώμη κάποιος εδώ πέρα μας τηλεφωνεί, μιλήσατε για μια ασφαλέστερη Ευρώπη, αναφέρατε τη διαδικασία της Οκχόλμης, πράγματι εδώ πέρα ανακύπτουν κάποιες δήματα ασφάλειας. Δεν αναφέρατε ρητός ε, την ε, ενεργειακή ασφάλεια που σχετίζεται νομίζω με τη στρατηγική της Βαλτικής την οποία αναφέρατε και άρα ερχόμαστε στο ρόλο της Ρωσίας. Αναρωτιέμαι πώς τα βλέπει όλα αυτά η Σουηδική Προεδρία. Το δεύτερο και τρίτο ερώτημα μου είναι πιο τεχνικά. Αυτή τη στιγμή πώς βλέπει η Σουηδική Προεδρία τη μελλοντική σχέση μεταξύ του μόνιμου Προέδρου του Συμβουλίου και του Πρωθυπουργού της χώρας που θα έχει την Προεδρία του Συμβουλίου. Και εδώ πέρα να συμπληρώσω το ερώτημα του κυρίου Νταφ. Όταν σκεφτόμαστε το πρόσωπο του μόνιμου πρόεδρου. Υπάρχει μήπως κάποια προτίμηση για κάποιον από ένα μικρό κράτος έναντι κάποιο από μια μεγάλη χώρα. Και τρίτο τεχνικό ερώτημα, ποιος είναι ο μηχανισμός, εάν υπάρχει, που στείνεται για να περάσουμε από την μία αυτή τριπλή προεδρία στην επόμενη. Για... Και αναρωτιέμαι γιατί η Ουγγαρία θα έχει το, το τέλος, αν θέλετε, της τριπλής προεδρίας θα ακολουθεί στην δική σας τριπλή προεδρία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο συνάδελφος Χέφνερ έχει το λόγο. Ja, auch von meiner Seite ein herzliches ναι και από μένα ένα καλώς ήρθατε στην κυρία Υπουργό και σας ευχαριστώ. Μια πρώτη παρατήρηση. Η εντύπωση μου είναι και νομίζω και των περισσότερων συναδέλφων πως η Ευρώπη ε, βρίσκεται σε μια δύσκολη διαδικασία και είναι πολύ ευτυχή συγκυρία ότι έχουμε Σουηδική Προεδρία. Θα ήθελα τώρα να θέσω δύο ερωτήματα. Το πρώτο αφορά την ε, εκλογή της, ε, προσεχής, της προσεχούς ε, με Κομισιόν και του Πρόεδρου της. Εδώ πέρα πολλοί συναδελφοί και ομάδα μας θεωρούν πως η Ευρώπη μπορεί να, να βρει καλύτερα και αξίζει καλύτερα από, τους, από τον υποψήφιο τον κύριο Μπαρόζο. Το ερώτημά μου είναι κατά την άποψή σας η απονομική σκοπιά το να μην έχουμε ενιαία εκλογή, δηλαδή το ότι εκλέγουμε τον πρόεδρο με τη μία συνθήκη και την υπόλοιπη κομισιόν με μία άλλη ε, συνθήκη. Τι εντύπωση δίνουμε δηλαδή στους πολίτες εμείς ως ε, θεσμικά όργανα. Δεύτερο ερώτημα αναφέρατε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα. Πρώτα απ' όλα την εμπιστοσύνη των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση που πρέπει να ενισχυθεί και το δεύτερο ήταν το ότι όταν και αν τεθεί ενισχύει η συνθήκη της Λισαβόνας θα καταβάλλεται κάθε ε, προσπάθεια για να ισχύσουν αμέσως το όσο αναφέρονται εκεί πέρα. Ε, εμένα μου φαίνεται σημαντικό το εξής. Οι πολίτες της Ευρώπης, τα κράτη-μέλη σήμερα έχουν τη δυνατότητα να εκφραστούν στην ε, πολιτική άμεσα και έμεσα. Και γι' αυτό νομίζω θα είναι σημαντικό, ειδικά επειδή η απόφαση λαμβάνεται αρκετά μακριά από τους πολίτες να μπορούν να εκφράζονται και υπάρχει ακριβώς αυτό το μέσο συνθήκης Λισαβόνας δηλαδή η πρωτοβουλία των πολιτών να μπορέσουν να ξεκινήσουν μια πρωτοβουλία για να ξεκινήσει μετά να ασχολείται η Κομισιόν με αυτό το θέμα. Το ερώτημά μου είναι τι θα κάνει η Σουηδική Προεδρία, πώς έχει ήδη ξεκινήσει έτσι ώστε να μπορέσει να κινηθεί αυτή η διαδικασία άμεσα μετά την ε, επικύρωση όπως ελπίζουμε της ε, συνθήκης γιατί έχει περάσει αρκετός χρόνος και θα μπορούσαμε λογικά να έχουμε κάνει κάτι, να έχετε κάνει εσείς κάτι προς αυτή την κατεύθυνση, δεν ξέρω είναι τόσο δύσκολο εδώ πέρα να έχουμε κάποιες προτάσεις για συγκεκριμένη εφαρμογή αυτής της διάταξης. Ε, Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σέντεργκάρντ έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Υπουργέ, κυρία Μάλμστρομ, που παρεμβήκατε σήμερα το πρωί εδώ. Θα ήθελα να σας υποβάλω τρεις ερωτήσεις. Η πρώτη αφορά την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Καρλς στη Γερμανία. Έγινε μία εις βάθος συζήτηση και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι πώς το συνταγματικό δικαστήριο αποφαίνεται σε σχέση με την υπεροχή του κοινοτικού δικαίου. Έγινε μια συζήτηση για το κατά πόσο η απόφαση του συνταγματικού δικαστηρίου είναι ένα καθαρά γερμανικό ζήτημα, ενδογερμανικό ή κατά πόσο έχει επιπτώσει στο κοινοτικό δίκαιο και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το δεύτερο ερώτημα, κυρία Μάλμστρεμ, σχετίζεται με το θέμα της ε, χαμηλής ε, του, του γεγονότος ότι υπήρξε πολύ χαμηλό ποσοστό συμμετοχής στις εκλογές. Δεν ξέρω κατά πόσο θα πρέπει να μας απασχολήσει και μας είχε απασχολήσει στην πρώτη τελευταία συνεδρίαση, όπως γνωρίζετε, κατά τη λήξη της ε, προηγούμενης θητείας σε σχέση με το, το, το θέμα των πόρων του 2007. Ξέρω ότι η Σουηδία θεωρεί πρώτη της σημασίας το θέμα του ότι όλα πρέπει να έχουν ένα ανοιχτό χαρακτήρα, δημόσιο χαρακτήρα. Και τι γνώμη έχετε για τους λογαριασμούς του 2007. Η Σουηδική Προεδρία θα, θέλει θα ήθελε να έχουμε όλες τις πληροφορίες για μια λογοδοσία του Συμβουλίου γιατί πολλές φορές ζητάμε πληροφορίες από το Συμβουλίο και πρέπει να εγκρίνουμε τους λογαριασμούς, αλλά δεν υπάρχει διαφάνεια. Το δεύτερο ζήτημα σχετίζεται με τη χαμηλή συμμετοχή στις ευρωεκλογέ. Και αυτό σχετίζεται και με τον κοινωνικό ιστό. Εσείς προέρχεστε από τη Σουηδία, όπου, είχα, όπου υπήρχε και η απόφαση Βάξχολμ. Το ΔΕΚ αποφάνθηκε ότι δεν είναι αποδεκτό να καταβάλλονται χαμηλότερα ημερομίσθια στους Πολωνούς εργαζόμενους, διότι στη Δανία οι Πολωνοί θεωρούνται πολίτες δεύτερης κατηγορίας και τους καταβάλλονται πολύ χαμηλότερα ημερομίσθια σε σχέση με τους Δανούς. Ε, μιλάμε για ευρωπαϊκή συνεργασία και πολλές φορές πολίτες άλλων ε, εθνικοτήτων Λαμβάνουμε ακόμα χαμηλότερα ημερομίσθια. Ξέρετε την απόφαση Βάξχολμ του ΔΕΚ. Ποια είναι η γνώμη της Σουηδικής Προεδρίας. Πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι να εγγυθούμε την απαληφή του κοινωνικού ντάμπινγκ έτσι ώστε να, να μην καταβάλλονται πλέον χαμηλότερα ημερομίσθια για άλλους Ευρωπαίους πολίτες στη χώρα εργασίας. Ο συνάδελφος Σαλάτο έχει το λόγο. Πρόεδρε, θα ήθελα να εκφράσω ορισμένες σκέψεις σε σχέση με την χθεσινή και τη σημερινή συζήτηση. Νομίζω ότι υπάρχουν δύο επιχειρήματα τα οποία είναι αλληλένδετα. Η συνθήκη της Λισαβόνας και η υψηλή αποχή στις ευρωεκλογές. Ως προς τη συνθήκη της Λισαβόνας δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για όποιον ε, γνωρίζει τα πολιτικά δρόμενα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θα πρέπει να προβούμε στην πραγμάτωση, της, ε, την υλοποίηση της συνθήκης της Λισαβόνας, έτσι ώστε η Ευρώπη να είναι πιο κοντά στους πολίτες. Εάν μπορώ να εκφράσω ειλικρινά την άποψή μου. Ε, δεν νομίζω ότι αυτό θα είναι και τόσο εύκολο. Θα είναι δηλαδή δυσεπίλητο και για το παρόν και για το μέλλον. Διότι είμαι πεπισμένος και αυτό δεν είναι μόνο προσωπική άποψη, αλλά έχει επιπτώσεις και στην ε, υψηλή αποχή στις ευρωεκλογέ, ότι με βάση τα ευρωπαϊκά συμφραζόμενα υπάρχουν μεγάλες δυνάμεις που δεν βλέπουν με καλό μάτι την μεγαλύτερη συμμετοχή στα πολιτικά κοινοβουλευτικά δρόμενα. Ε, προτιμούν, ε, αυτό το καταδεικνύουν και οι έρευνες. Ε, ας δούμε τις γραφειοκρατικές επιπτώσεις που υπάρχουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και που δυσχεραίνουν την δράση των Ευρωπαίων πολιτών. Αν μιλάμε λοιπόν για τη συνθήκη της Λισαβόνας και αν θεωρούμε τη συνθήκη πανάκια, αυτό νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα αισιόδοξο και άγωνο. Υπάρχει όμως και το άλλο ζήτημα, το θέμα της συμμετοχής των πολιτών, δύναμη της συνθήκης της ε, Λισαβόνας. Αλλά αν δεν υπάρχει μεγαλύτερη δημοσιοποίηση της λειτουργίας του Ευρωπαϊ... της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Επιτροπής, δεν θα γίνει κάτι τέτοιο. Εγώ μιλώ για τη χώρα μου, στην Ιταλία. Το 80% δεν γνωρίζουν ότι η νομοθετική ε, διαργασία γίνεται στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ μιλώ για τη χώρα μου. Δεν θέλω να μιλήσω για άλλες. Ο Ευρωβουλευτής ε, θεωρείται από τους εθνικούς βουλευτές ότι είναι ένας ελέφαντας ο οποίος μεταβαίνει στο κημητήριο ελεφάντων κάθε μήνα. Αυτή η θεώρηση υπάρχει ως προς το ρόλο μας και ότι ο Ευρωβουλευτής ε, πληρώνεται πολύ και υπερβολικά και έπρεπε να εξηγήσω στους περισσότερους φίλους ότι δεν ισχύει αυτό που αναφέρεται ως προς τους ε, ευρωπαϊκούς μισθούς. Αυτό σημαίνει ότι σε κάθε χώρα υπάρχουν ε, δίκτυα πληροφοριών, αρχίζοντας από τον τύπο, που επειδή ακριβώς διέπονται και χειραγωγούνται από μεγάλες δυνάμεις, δεν προβαίνουν στη σωστή πληροφόρηση, όπως κάνουμε εμείς μέσω Ευρωκοινοβουλίου. Θα ήταν λοιπόν σκόπιμο, αναμένοντας την υλοποίηση της συνθήκης της Λισαβόνας, τα αρμόδια ε, όργανα, οι διασκέψεις να προωθήσουν αυτό το δίκτυο πληροφοριών έτσι ώστε οι πολίτες να αναγνωρίσουν πόσο σημαντική είναι η ζωή και η δράση του Ευρωκοινοβουλίου για τα δικά του συμφέροντα. για το έργο αυτό το οποίο θα πρέπει να γίνει γνωστό. Έτσι ώστε να πείσουμε τους πολίτες για το ρόλο μας. Θα ήθελα λοιπόν να κάνω μία έκκληση στη Σουηδική Προεδρία και στην Υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων να εξεύρει λύσεις μεγαλύτερης επίπτωσης στους ε, μηχανισμούς πληροφόρησης. Δεν ξέρω τι συμβαίνει σε άλλες χώρες, δεν νομίζω όμως ότι διαφέρει η κατάσταση από τη δική μας. Αν διαβάσετε μέρος του ημερήσιου τύπου, το βλέπετε αυτό. Η τηλεόραση προβλέπει ένα πρόγραμμα ημιόρου κάθε Σάββατο για ευρωπαϊκά ζητήματα και τίποτα άλλο. Και εάν δώσουμε μία όθηση στα ΜΜΕ που την χάνουν κρατικής υποστήριξης και κρατικής χρηματοδότησης, Εάν λοιπόν επιβάλλουμε μία μεγαλύτερη και καλύτερη πληροφόρηση, τότε θα έχουμε κάνει κάτι το πολύ θετικό πέρα από τη συνθήκη της Λισαβόνας και θα είμαστε σε θέση να συνεισφέρουμε ουσιοδός στις ε, συζητήσεις και στην πληροφόρηση αυτή, κάτι το οποίο είναι ύψη της σημασίας για την ανάπτυξη της Υπήρου μας. Ευχαριστώ. Τελευταίος ομιλητής, ο Σνάδος Κρασκόφσκι. <clears throat> Υπουργέ, θα ήθελα να σας υποβάλω μια ειδική ερώτηση. σας ερώτησαν πού βρισκόμαστε όσον αφορά αυτή την εξωτερική υπηρεσία της Κομισιόν. Θα ήθελα να είμαι πιο ειδικό. Ποια είναι η δική σας προσέγγιση. Διότι η πρώτη προσέγγιση πριν από το δημοψήφισμα ήταν να παρουσιάζονται αυτά τα επίσημα τα δελτία. Έχω την εντύπωση λοιπόν ότι πολλές κυβερνήσεις πανικοβλήθηκαν, διότι συνειδητοποίησαν ποιες θα είναι οι άμεσες επιπτώσεις από τη συνέχιση της Λισαβόνας, διότι υπάρχουν δύσκολα θέματα. Δηλαδή, τι θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει, πώς θα λυθούν τα οικονομικά θέματα, ποιος θα είναι ο νέος ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όταν θα συσταθεί αυτή η εξωτερική υπηρεσία. Το ερώτημα ξέρω ότι είναι πάρα πολύ ευαίσθητο, αλλά ερωτώ, ποια νομίζετε θα είναι η δική σας προσέγγιση, έχετε συγκεκριμένες προτάσεις όταν ολοκληρωθεί το δεύτερο ε, δημοψήφισμα στην Ιρλανδία και ελπίζουμε ότι καταλήξει στα αποτελέσματα που αναμένουμε. Θα αποστείλετε και πάλι ερωτηματολόγια ή θα υποβάλλετε επιτάπητος συγκεκριμένες προτάσεις. Επίσης, έχετε άτυπες επαφές με άλλες κυβερνήσεις ή έχουν παγώσει τα πάντα σε σχέση με αυτό το θέμα. Ξέρω, επαναλαμβάνω, ότι είναι δύσκολο το θέμα αυτό, αλλά θα ήθελα να μας πείτε ποια είναι η δική σας απάντηση και ξέρω ότι εσείς είστε υπέρ της διαφάνειας σε τέτοιους θέματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι έχουμε υλικό για σκέψη, τροφή για σκέψη και εγώ θα ήθελα να προσθέσω ε, ένα ερώτημα προς την Υπουργό αν και κατανοώ ότι δεν μπορεί να τύχει άμεση απάντηση, όπως πολλές από τις ερωτήσεις που υποβλήθηκαν. Θα ήθελα όμως να εκφράσω την άποψή μου μέσα στα πλαίσια ενός σκεπτικού για τις ε, μελλοντικές μας εργασίες. Μέχρι ποιου σημείου το θέμα της ε, μετανάστευσης απασχολεί την ευρωπαϊκή συλλογική συνείδηση. Διότι ορισμένες χώρες αντιμετωπίσουν μια κατάσταση κρίση, όπως η δική μου. Και τη στιγμή που μιλάμε για ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που επικεντρώνει το πρόγραμμά της στα ανθρώπινα δικαιώματα, στα δικαιώματα των πιο φτωχών, στην ανάπτυξη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα ιδεώδες το οποίο βεβαίως ε, κινείται και στα πλαίσια καταπολέμησης και πάταξης της εγκληματικότητας όταν μιλάμε για πρόσωπα που υπόκεινται σε, σε καταστάσεις βίας. Θεωρούμε ότι αυτό αποτελεί το επίκεντρο της σκέψης μας. Θα το αντιμετωπίσει η Ευρώπη χωρίς να αφήσει το θέμα στα μεμονωμένα κράτη-μέλη. Σας ευχαριστούμε πολύ και αναμένουμε τις απαντήσεις σας. Ευχαριστώ κύριε και κύριοι. Νομίζω πως ε, κάθε μία ερώτηση είναι σεμινάριο από μόνη της, γιατί είναι δύσκολες και πολυπλοκές, αλλά θα προσπαθήσω να απαντήσω σύντομα σε όλες. Ε, ξεκινώντας από τον φίλο μου τον κύριο Μαντεστε Βίγκο. Θίξατε ένα ζήτημα που ανέφεραν και άλλοι συναδελφοί, τον είπα το εκπρόσωπο και την υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Για τον είπα το εκπρόσωπο και το πώς θα επικοινωνήσουμε με το Κοινοβούλιο. Είναι σημαντικό αυτό το ζήτημα. Πράγματι την Παρασκευή θα, συναντήσω με το, θα συναντηθώ με, με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, τον κύριο Μπούζεκ. Ναι, αυτή την Παρασκευή για αυτό το θέμα και για πολλά άλλα για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να επικοινωνούμε, να συνεργαζόμαστε όσο το δυνατόν πιο ομαλά. Ξέρω πως σας απασχολεί αυτό το ζήτημα, απασχολεί και εμάς για να δούμε την διαδικασία όσον αφορά την υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Στόχος μας είναι αν όλα κυλήσουν ομαλά και επικυρωθεί η συνθήκη της Λισαβόνας, εάν λέω, τέλος Οκτωβρίου στο Συμβούλιο να αποφασίσουμε όλα αυτά τα θεσμικά ζητήματα, να καταλήξουμε σε έναν κατάλογο επιτρόπων που θα σταλεί να ορίσουμε, είπα το εκπρόσωπο, και να ορίσουμε και πρόεδρο του Συμβουλίου. Επίσης ελπίζουμε πως θα μπορέσουμε να ευθύσουμε ένα πλαίσιο αρκετά χαλαρό για την υπηρεσία εξωτερικής δράσης υπό την προϋπόθεση πως ε, η ίδια, ο ίδιος ο ύπαθος εκπρόσωπος θα επανέλθει στο Συμβούλιο και βεβαίως θα έχει και διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αυτό το θέμα. Κάποια από τα άλλα ζητήματα που έθιξαν οι λοιποί συναδελφοί αντιμετωπίστηκαν επί Σλοβενικής ε, Προεδρίας, κάτι το οποίο μας ε, διευκολύνει πάρα πολύ. Συμφωνώ πως ε, ήταν πολύ δύσκολα και ευαίσθητα αυτά τα ζητήματα και δεν τα είχαν επεξεργαστεί τελείως όλα τα κράτη-μέλη π.χ. για το πώς θα ορίζονται αυτοί οι υπάλληλοι, το καθεστώς τους, ε, το πώς θα χρηματοδοτείται η υπηρεσία. Αυτά δεν έχουν ξεκαθαρίσει ακόμα και από σεβασμό και για την απόφαση του Ιρλανδικού λαού δεν μπορούμε ακόμα να καταθέσουμε πιο συγκεκριμένες προτάσεις, αλλά έχει υπάρξει μια προεργασία από τη Σλοβενική Προεδρία και βεβαίως οι συζητήσεις ε, συνεχίζονταν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, οπότε θα έχουμε Εκτεταμένε συζητήσεις για να καταλήξουμε όταν έχουμε κάποιο οριστικό αποτέλεσμα και θα έχουμε συγκεκριμένες προτάσει όταν ακούσουμε και όλες τις σχετικές απόψεις. Όπως σα είπα κάποια προεργασία έχει γίνει αλλά βεβαίω έπρεπε να αναμένουμε και την απόφαση της Ιρλανδίας και δεν θέλουμε να προδικάσουμε το αποτέλεσμα. Με ρωτήσατε για κάποια άλλα προβλήματα πέραν της επικύρωσης στην Ιρλανδία. Προφανώς μας λείπει ακόμα η υπογραφή του Πολωνού Προέδρου. Γνωρίζουμε πως η διαδικασία στην Γερμανία έχει ένα χρόνο διάγραμμα. Οι Γερμανοί συνάδελφοί μας λένε πως θα οριστικοποιηθεί αυτό κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου πριν από το δημοψήφισμα στην Ιρλανδία και μετά έχουμε και διαφορετικές διαδικασίες στην Πράγα που δεν ξέρουμε πότε θα ολοκληρωθούν. Απλά θα ήθελα να σα υπενθυμίσω, το γνωρίζετε βεβαίω, πω όλε οι χώρες έχουν δεσμευτεί να καταβάλουν κάθε προσπάθεια έτσι ώστε να τεθεί ενισχύ η συνθήκη και αν και οι στην Πράγα έχουν επικυρώσει με επαρκή πλειοψηφία την συνθήκη, οπότε ελπίζουμε πως θα λυθούν αυτά τα ζητήματα κατά τη διάρκεια του φθινοπόρου, αλλά όλες οι χώρες πρέπει να ολοκληρώσουν τη διαδικασία επικύρωσης της συνθήκης και αν δεν γίνει αυτό δεν θα ισχύσει η συνθήκη της Λισαγώνας. Οπότε ελπίζουμε πως θα λυθούν αυτά τα ζητήματα. Έχουμε βεβαίω και το, το δημοψήφισμα της Ιρλανδίας στις 2 Οκτωβρίου. Κύριε Χάγκη, εσείς και κάποια άλλη ρωτήσατε για τον πρόεδρο της Κομισιόν γιατί να οριστεί τώρα. Θεωρούμε πως αντιμετωπίζουμε εξαιρετικές περιστάσεις. Έχουμε την μεγάλη οικονομική κρίση και το θέμα του κλίματος, ε, ζητήματα που απαιτούν έναν ηγετικό ρόλο της Ευρώπης ε, σε παγκόσμια κλίμακα. Ομόφωνα το Συμβούλιο όρισε τον κύριο Μπαρός ως υποψήφιο, κυκλοφορούσε βέβαια στο όνομά του και πριν από τις ευρωεκλογές, είναι γνωστός υπήρχε μια κεντροδεξιά πλειοψηφία που προέκυψε από τις ε, ευρωεκλογές. Το Συμβούλιο αποφάσισε πως ακόμα και χωρίς τη συνθήκη της Λισαβόνας εμείς θέλαμε τον κύριο Μπάρος ως πρόεδρο και θεωρούν πως είναι σημαντικό με την οικονομική κρίση όλα αυτά που πρέπει να γίνουν με την κλιματική κρίση το διοσυναριακό έγκλημα, το ζήτημα της μετανάστευσης που ανέφερε ο Πρόεδρος και στο οποίο θα επανέλθω πρέπει να ε, έχουμε αυτά αποτελέσματα για τους πολίτες μας σε όλα αυτά. Και εδώ πέρα έρχομαι και στο τρίτο ερώτημά σα. Γιατί δεν ψηφίζουν στι ευρωεκλογέ οι άνθρωποι, γιατί δεν του απασχολούν τα ευρωπαϊκά ζητήματα. Ίσως γιατί εμεί και εγώ, γιατί είμαι και πολιτική, πολιτικός επιστήμον, Ίσως ε, ασχολούμαστε πάρα πολύ με τα θεσμικά ζητήματα και όχι με τα καθημερινά ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες. Τους απασχολεί το αν έχουν δουλειά, τους απασχολεί η κλιματική αλλαγή, τους απασχολεί το διοσυναριακό έγκλημα. Και πρέπει να έχουμε αποτελέσματα. Βεβαίω, για αυτά χρειαζόμαστε για να γίνουν με διαφανή δημοκρατικό και νόμιμο τρόπο τα κατάλληλα θεσμικά όργανα. Αυτό είναι το καλύτερο το οποίο μπορούμε να κάνουμε λοιπόν για αυτούς, να τους δείξουμε πως είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε ηγετικό ρόλο και να έχουμε αποτελέσματα. Αντιλαμβάνουμε βεβαίω πως ε, ενώ μόλι είχε εκλεγεί τον Ιούλιο το Κοινοβούλιο δεν ήταν σε θέση να εκλέξει πρόεδρο. Έπρεπε να συσταθεί σε σώμα ή επιτροπές κτλ. Ελπίζω λοιπόν να μπορέσετε να εγκρίνετε τώρα τον κύριο Παρόσο για να βοηθήσετε και το Συμβούλιο και την Κομισιόν στο σημαντικό έργο που μας περιμένει. Τώρα για τη στρατηγική της Λισαβόνας. Ναι, είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα και η Σουηδική Προεδρία το έχει πολύ ψηλά στις προτεραιότητες της. Σε όλους τους σχηματισμούς του Συμβουλίου θα συζητηθεί που είχαμε επιτυχίες, που όχι, κάποια τμήματα ήταν πολύ πιο επιτυχή από άλλα, τι μπορούμε να κρατήσουμε για το μέλλον δεν είναι ένα μέσο για να βγούμε μόνο από την τωρινή κρίση, είναι ένα μακροπρόθεσμο μέσο για να αποκαταστήσουμε την αξιοπιστία των χρηματαγορών και την ε, φόρο και βιώσιμη ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Και βεβαίως θα πρέπει να συζητήσουμε και το πώς χρησιμοποιούμε τον προϋπολογισμό μας. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να το εξάσουμε όσο πιο αναλυτικά γίνεται. Θα έχουμε πολλές διασκέψεις επί Σουηδικής Προεδρίας και το Μάρτιο η Ισπανική Προεδρία, όπως γνωρίζετε, σκοπεύει να το κλείσει αυτό το θέμα και πιθανώς να βγάλει κάποια συμπεράσματα και μια απόφαση στην ε, Σύνοδο Κορφής του Μαρτίου. Ο πρόεδρος του Συμβουλίου τώρα. Αναφέρεται στην συνθήκη ο ρόλος του ή ρόλος της Ε, ίσως δεν θα πρέπει αυτή τη στιγμή να προσπαθήσουμε να ερμηνεύσουμε τη συνθήκη. Η συνθήκη υπάρχει, αναφέρεται και ο ρόλος όταν τεθεί ενισχύ θα πρέπει να συζητήσουμε και τις διάφορες απόψεις των κρατών μελών και του Κοινοβουλίου για τον ρόλο και της ε, εναλλασσόμενης ε, Προεδρίας και πώς θα λειτουργήσει το, το ζήτημα. Είναι κάπως πρόωρο αυτή τη στιγμή να μπούμε σε λεπτομέρειες. Αυτή τη στιγμή θα έλεγα πως ακούμε όλα τα κρατημέλη και τα θεσμικά όργανα και τελικά θα κάνουμε κάποιες ε, προτάσεις. Όπως είπα τον Οκτώβριο, εάν ε, προχωρήσουν ομαλά οι διαδικασίες επικύρωσης, η Σουηδική Προεδρία δεν έχει κάποιο ρόλο στο Ιρλανδικό Δημοψήφισμα έχουμε επιδείξει μια προθυμία έναντι της Ιρλανδικής κυβέρνησης να τους στηρίξουμε αν θέλουν. Αλλά δεν ε, έχει γίνει κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή. Παρακολουθούμε βεβαίω την συζήτηση στην Ιρλανδία περί Τούρκων αγροτών και λοιπόν και στις διάφορες ε, ιστοσελίδες γίνονται αυτές οι συζητήσεις. Είναι πολύ έντονη συζήτηση, ελπίζω να υπάρχει και μεγάλη συμμετοχή και θετικό αποτέλεσμα. Αλλά δεν θεωρούμε εμεί ω Ειδική Προεδρία καθήκον μας να παρέμβουμε. Και σας ευχαριστώ και για την πρόταση σας για μια τελετή. Θα το εξετάσουμε. Όπως είπε ο κύριος Φόξ. Ναι, για τον είπα το εκπρόσωπο ακόμα εξετάζουμε προτάσεις. Δεν έχω ακούσει τη Βρετανική πρόταση εγώ έχω ακούσει εκτός από αυτήν άλλα 15-20 ονόματα που κυκλοφορούν αν διαβάζει κανείς τις εφημερίδες, φήμες και διάφορα. Ακούμε όλα αυτά τα ονόματα, αλλά η εμπειρία μας λέει πως όσο πιο κοντά πλησιάζουμε στην διαδικασία τόσο πιο πολλά ονόματα θα ακουστούν. Είναι πολύ νωρί να ορίσουμε ακόμα κάποιον σε μια δουλειά, σε μια θέση η οποία δεν υφίσταται. Δεν είναι ακόμα ενισχύει συνθήκη. Δεν θέλω λοιπόν να κάνω εικασίες. Με ρωτήσατε για τη Βυρμανία. Συμφωνώ με την ανησυχία σας. Γενικά τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι προτεραιότητα τη Σουηδική Προεδρίας. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο έχει συζητήσει αρκετές φορές ε, το ζήτημα της Βυρμανίας και κατά τη διάρκεια της ε, δίκης καταδίκης και σύλληψης κυρίας ε, Σουνκή είχαμε επανειλημμένα διαμαρτυρηθεί και αποφασίσαμε τον Αύγουστο να επιβάλλουμε και άλλες ε, κυρώσεις στη Γερμανία. Είναι δύσκολο να έρθουμε σε επαφή με αυτό το, το καθεστώς, αλλά συμφωνώ με τις ανησυχίες σας κύριε Φόξ. Κύριε Σεφλίν, για τη Ρωσία. σκοπεύουμε να γίνει μια σύνοδος κορυφής με την Ρωσία το φθινόπωρο. Θα επανέλθω με λεπτομέρειες. Είναι βεβαίως μια σημαντική γείτονας. Διαπραγματευόμαστε μια νέα συμφωνία. Βεβαίως η ενεργειακή ασφάλεια θα είναι στα θέματα που θα συζητηθούν μαζί με άλλα ζητήματα και η γενικότερη ασφάλεια αλλά και γενικώ στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αλλά και ειδικά στο πλαίσιο των σχέσεων με την Ρωσία και για τι πρωτοβουλίε πολιτών. Ήταν δικό σα αυτό το ερώτημα, όχι ο κ. Σέφνερ. Ναι. Και η κυρία Κάφμαν νομίζω είχε συντάξει μία έκθεση στην Επιτροπή σας πέρσι με προτάσεις για το πώς θα πρέπει να προχωρήσει αυτό το ζήτημα. Εμείς αναμένουμε από την Κομισιόν να επανέλθει το μόνο δυνατόν μετά την θέση ενισχύ τη ε, συνθήκη. για με συγκεκριμένες για το πώς θα εφαρμοστεί ε, άμεσα αυτό, γιατί είναι πραγματικά κάτι πολύ σημαντικό, ένα πολύ σημαντικό τμήμα της συνθήκης που αφορά άμεσα του πολίτε. Ναι, και Σέφλιν, εσείς ρωτήσατε για τις ε, τριπλές αυτές ε, προεδρίες. Είχαμε πολύ καλή συνεργασία με Τσέχους και Γάλλους πριν και πριν από την Γαλλική Προεδρία και ήταν πάρα πολύ χρήσιμο αυτό και εμείς ως Σουηδική Προεδρία φροντίσαμε να εμπλέξουμε και την επόμενη τρίπλη Προεδρία, το επόμενο τρίο. Εγώ έχω συναντηθεί και είχαμε και γευματεργασίας ε, και με την επερχόμενη τριπλή προεδρία Ουγγαρία, Ισπανία, Βέλγιο και οι έξι συνάδελφοι αρκετές φορές για να συντονίσουμε την όλη διαδικασία, το ποια είναι τα ζητήματα στην ατζέντα και πολύ συγκεκριμένα για την ε, Ισπανική Προεδρία που ακολουθεί. Έχουμε καθημερινές επαφές ε, στις ομάδες εργασίας, οπότε ελπίζουμε πως η μετάβαση να γίνει όμαλα και βεβαίως η εμπειρία αυτή της ε, τριπλής Προεδρίας μας βοήθησε πάρα πολύ, βοήθησε να εγγυηθούμε μια συνέχεια και μια σταθερότητα στο έργο της Ένωσης. Κύριε Σαντεγκάρτ, στο πλαίσιο του Συμβουλίου δεν ε, έχουμε συζητήσει την απόφαση του Γερμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου. Βεβαίως όλοι παρακολουθήσαμε με μεγάλη προσοχή την εξέλιξη αυτή. Κάθε χώρα έχει διαφορετικές διαδικασίες. Εσεί στη Δανία και εμείς Σουηδία έχουμε πολύ ισχυρό κοινοβουλευτικό έλεγχο επί του, του Συμβουλίου. Η κάθε χώρα έχει διαφορετικούς μηχανισμούς. Ε, η Γερμανία έχει τους δικού τη. Εμείς δεν θεωρούμε πως υπάρχει κάποιο λόγο να παρέμβουμε σε αυτό. Το Συνταγματικό Δικαστήριο είπε επίση πω δεν αντιβαίνει στο γερμανικό σύνταγμα η Σύνθηκη Λισαβόνας, απλά πρότεινε κάποιες αλλαγές και στην Ομοσπονδιακή Βουλή και στο Ομοσπονδιακό Συμβούλιο. Ξέρω πως είστε εσείς ο υπεύθυνο ο εισηγητής. Μπορείτε να έρθετε σε επαφή είτε με μένα είτε με έναν συνάδελφό μου για να δούμε αν υπάρχουν κάποιες ασάφειες. για την απόφαση Βάξχολμ. Ίσως δίνουμε διαφορετική ερμηνεία. Δεν είναι πράσινο φως για κοινωνικό ντάμπινγκ. Θεωρούμε πως πρέπει να γίνουν κάποιες ε, αλλαγές, εμεί θεωρούμε, στην Σουηδία. Υπάρχουν διαφορετικές περιπτώσεις στην Ευρώπη. Υπάρχει μια ομάδα υψηλού επίπεδου τους κοινωνικούς εταίρους, να δούμε πώς θα ερμηνεύσουμε την ε, οδηγία περί αποσπάσεως ε, εργαζομένων για να μπορέσουμε να, να συμμορφωθούμε με την απόφαση. Οπότε το εξετάζουμε και στο ευρωπαϊκό και στο σουηδικό επίπεδο. Και τα σκόψη νομίζω ότι απάντησα. Ελπίζουμε να έχουμε μια απόφαση πλαίσιο τον Οκτώβριο και ο νέος ύπατος εκπρόσωπος, εάν οριστεί με την συνθήκη της Λισαβόνας, θα επανέλθουμε μια πρόταση και θα πρέπει να συζητηθεί κατόπιν αυτή. Οπότε, κύριε Πρόεδρε, τέλος. Ναι, πράγματι η μετανάστευση είναι σημαντικό ζήτημα, απασχολεί πολλές ομάδες του Συμβουλίου, παρακολουθούμε τη συζήτηση που γίνεται στην Νότια Ευρώπη τις τελευταίες εβδομάδες, είναι πάντα ένα ζήτημα που απασχολεί, είναι στο πλαίσιο του προγράμματος Σοκχόλμης. είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα που δεν μπορεί να λυθεί σε μια συνεδρίαση του Συμβουλίου. Θα πρέπει όμως να δούμε και ποια είναι τα ωφέλη της μετανάστευσης, γιατί χρειαζόμαστε νόμιμη μετανάστευση και να λύσουμε και το δημογραφικό της Ευρώπης, αλλά να δούμε και πώς μπορούμε να βοηθηθούμε όταν μιλάμε για την παράνομη ε, μετανάστευση, για να αποφύγουμε και αυτές τις τραγωδίες και τον ανθρώπινο πόνο που είδαμε τους καλοκαιρινούς ε, μήνες. Οπότε σας διαβέω πως οπωσδήποτε θα επανέλθω σε αυτό το σημείο. Αυτά ελπίζω να απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις σας. Σας ευχαριστώ. Allora, io ringrazio... Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους όσους συμμετείχατε στη συζήτηση με ενδιαφέρουσες ερωτήσεις. Ευχαριστώ και την κυρία Μάλστρεμ που παρευρέθηκε εδώ μαζί μας. Σας ευχαριστώ για τις διεξοδικές σας απαντήσεις, αν και προϋποθέτουν μελλοντικές εργασίες. Γνωρίζουμε όμως ότι θα ασχοληθείτε εις βάθος με αυτά τα ζητήματα, έχετε δεσμηθεί και θα έρθετε εδώ πριν από το τέλος της ε, Προεδρίας και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά εξ ονόματος όλων.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 Μπορούμε να συνεχίσουμε με τις εργασίες μας. Μπορούμε να επεκταθούμε στο δεύτερο μέρος της συνεδρίασης εξετάζοντας τα άλλα σημεία της ημερήσιας διάταξης Υπενθυμίζω ότι η συνάντηση που είχαμε σήμερα με την ε, κυρία Μάλστρομ θα έχει και συνέχεια. Γιατί ο πρόεδρος Μπούζεκ θα παρευρεθεί εδώ την επόμενη Δευτέρα. Ελπίζω λοιπόν να καταστεί σαφές το ενδιαφέρον μας μέσα στα πλαίσια της συνεργασίας μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ιδιαίτερα στα πλαίσια των εργασιών της ΑΦΚΟ. Θα ήθελα τώρα να εξετάσουμε τα σημεία 8, 9 και 10 της ημερήσιας διάταξης που αφορούν τη γνωμοδότησή μας επί του προϋπολογισμού. Το προϋπολογισμός αφορά τον προϋπολογισμό μάλλον αυτής της Επιτροπής, λέει ο Πρόεδρος, αλλά και τον ε, προϋπολογισμό στην ολότητά του. Νομίζω ότι θα πρέπει να εξετάσουμε και τα δύο σημεία από κοινού, εξαιτίας της αιτιόδους συνάφειάς τους. Κατά την ε, προηγούμενη συνεδρίαση, με βάση τις υποδείξεις Σέπφλιν, μιλήσαμε για τροπολογίες. Αυτή τη στιγμή είναι 14 οι τροπολογίες. Έξι Σέπλιν, ε, έξι Μέσερ Σμιτ και ο κύριος Μέσερ Σμιτ μπορεί να έρθει εδώ. Πού είναι ο κύριος Μέσερ Σμιτ? Α, εντάξει. Όλοι οι αντιπρόεδροι, εν πάση περιπτώσει, μπορούν να έρθουν εδώ στα έδρανα. Δεν χρειάζεται και τόση ταπεινοφροσύνη, λέει ο πρόεδρος. Λοιπόν, έχουμε έξι τροπολογίες ε, Σεφλίν, έξι Messerschmitt, Λάμπερτ και Γκουαλτιέρι. Θα πρότεινα καταρχήν ο συντάκτης γνωμοδότησης να εκφράσει την απόψή του, μετά να γίνει αιτιολόγηση και αν θεωρεί ο εισήγητης θα ανταπαντήσει και θα περάσουμε στην ψηφοφορία. Εν πάση περιπτώσει θα ήταν σκόπιμο ο κύριος Σέπφλιν να εκφραστεί. Ευχαριστώ. Συμφωνώ ότι είχαμε μία διεξοδική συζήτηση την τελευταία φορά και δεν θα ήθελα να καταχραστώ του χρόνου σας δεν θα παρουσιάσω τις ε, ε, τροπολογίες μου. Σχετίζονται με την ε, στρατηγική ε, επικοινωνίας και πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει επικοινωνία με τους πολίτες και να έχουμε ένα set aside επ' αυτού. Πολλές τροπολογίες αντιτίθενται αυτό είναι σκόπιμο στα πλαίσια των δημοκρατικών διαδικασιών και αυτά θέλω να πω. Δεν θέλω να πω και κάτι άλλο. Θέλουμε να προωθήσουμε την Ευρώπη για τους πολίτες και για οποιασδήποτε περαιτέρω πληροφορίες είμαι σε θέση να, θα είμαι σε θέση να σας απαντήσω, ελπίζω. Ωραία θέλουν ε, όσοι υπέβαλαν τροπολογίες, οι υποβάλλοντες να ε, λάβουν το λόγο. Ο κύριος Μέσερ Σμιτ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι έχουμε ε, εμπειρική, ότι υπάρχει εμπειρική αιτιώδη συνάφεια σε σχέση με τα ποσά που διατέθηκαν και στην προεκλογική εκστρατεία και, την, ε, και το ποσοστό συμμετοχής που ήταν ιδιαίτερα απογοητευτικό. Γι' αυτό νομίζω ότι είναι αμφίσιμη η ε, διατύπωση του κειμένου ή πολλών κειμένων θα πρέπει να υποθέσουμε ότι θα εγκριθεί η συνθήκη της Λισαβόνας και γι' αυτό υπάβαλα και αυτές τις τροπολογίες, ελπίζω να τύχουν τις έγκριση της Επιτροπής. Ε, δεν θα ήθελα να παρέμβει κάποιος άλλος. Έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, έχω υπολογία στην ε, πρόταση γνωμοδότησης Απλώς υπάρχει ένα μικρό λάθος. Υπάρχει μέσα η λέξη ελευθερία όπως φαίνεται στο κείμενο, αλλά η σωστή λέξη είναι ευημερία. Είναι prosperity. Η σωστή λέξη. Αντί της ελευθερίας είναι η σωστή λέξη ευημερία. Ωραία. Εγώ ακούω στα Ιταλικά, λέει ο Πρόεδρος. Άκουσα την παρέμβαση στα Ιταλικά. Δεν ξέρω αν υπάρχει πρόβλημα μετάφρασης ή εάν το κείμενο είναι σωστό και που έγκυται το λάθος, λέει ο Πρόεδρος. Mr. President, the is... Το πρόβλημα είναι ότι αντί για τη λέξη ελευθερία η σωστή λέξη είναι ευημερία. Αντί για ελευθερία, ευημερία. Πρέγω. Σέφλιν. Πρόεδρε, θα ήθελα να πω ότι μπορώ να δεχτώ μια προφορική τροπολογία, όπως πρότεινε η κυρία Γιαννάκου την κατάλληλη στιγμή. Πρέγω, Νταφ. Θα ήθελα να θίξω το ζήτημα της τροπολογίας 6507. 6507 που αφορά την κοινωνία των πολιτών. Δηλαδή τον τόπο στις Βρυξέλλες, η πρόταση χρηματοδότησης ενός πιλωτικού προγράμματος για γραφεία για τις μη κυβερνητικέ που θα ασχοληθούν με την ε, κοινότητα πολιτών, τον οίκο της Ευρωπαϊκής Κοινωνίας των Πολιτών. Πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση, αλλά θα πρέπει να τύχει περαιτέρω σκέψης και θα πρέπει να συζητηθεί σε επίπεδο Επιτροπής. Γιατί για λόγους χρονισμού, timing, δεν ζητήσαμε τη γνωμοδότηση Επιτροπής. Θα πρότεινα λοιπόν να συμφωνήσουμε με την τροπολογία προς υπόμνηση pour mémoire αλλά να βγάλουμε το αριθμητικό στοιχείο των 350.000 ευρώ που υπάρχει στις πληρωμές και στις αναλήψεις. Δηλαδή να το αφήσουμε κενό. Δεν ζητάμε από την Επιτροπή Προϋπολογισμών να ψηφίσει επί ενός ποσού. Αλλά ζητούμε, την παρακινούμε μάλλον, να επανέλθει στο ζήτημα και να σκεφτεί την πρόταση ξανά, σε μεγαλύτερο βαθμό λεπτομερίας να σκεφτεί την πρόταση σε βάθος. Ε, ο εισηγητής κάτι θέλει να πει, παρατηρήσεις. Α, με συγχωρείτε, δεν σας είδα. Έχετε το λόγο. κολέγα. Έφνερ. Ja, ich möchte just zu dem von Andrew Duff angesprochenen Antrag kurz etwas sagen. Äh, ich denke, dass wir σχέση με αυτά τα οποία είπε ο κύριος Αυκύριε Κασάνη. Θα πρέπει να δούμε πώς η ευρωπαϊκή κοινωνία των πολιτών είναι κάτι το οποίο βλέπουν οι πολίτες. Πώς θα μπορέσουμε να ενεργήσουμε σωστά, διότι υπάρχουν διάφορα λόμπι, υπάρχουν διάφορες ε, που ενεργούν πιο εύκολα και υπάρχουν διάφορες ομάδες από την ε, κοινωνία των πολιτών που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στα πράγματα. Θα πρέπει λοιπόν το θέμα αυτό να εξεταστεί πιο διεξοδικά. Δεν νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να έχουμε ένα σφαιρικό ποσό στον προπολογισμό, αλλά να γίνει κάποια μελέτη για να δούμε με μεγαλύτερες λεπτομέρειες τι χρειάζεται και με ποιο τρόπο. Πιστεύω ότι μπορούμε να υποστηρίξουμε αυτή την ε, πρόταση και κάποιοι συνάδελφοι μπορεί να είναι απόντες, αλλά εγώ μπορώ να υποστηρίξω αυτή την ε, πρόταση που υπέβαλε ο κύριος Νταφ. Ευχαριστώ. Κύριος Χέπφεν. Ευχαριστώ πολύ. Ε, μπορώ να συμφωνήσω με αυτό το προσυπόμνηση που πρότεινε ο κύριος Νταφ. Χρειαζόμαστε όμως περαιτέρω μελέτες και σωστά ήταν αυτά τα οποία είπε ο Άντριου. Να συζητήσουμε περαιτέρω το θέμα ε, με την Κομισιόν. Μπορώ λοιπόν να δεχθώ αυτή την συμβαστική λύση που προτείνει και το προσυπόμνηση, το PM. Ναι. Απλώς θέλω να πω ότι η τροπολογία που προτείνουμε κινείται προς την κατεύθυνση των προτάσεων του εισηγητή. Είναι μια αιτιολογημένη τροπολογία που ενισχύει το κείμενο του εισηγητή, όπως κατέδειξε και η χθεσινή συζήτηση θα πρέπει να προωθήσουμε μία ποιοτική πολιτική συζήτηση με βάση τα ευρωπαϊκά πολιτισμικά δεδομένα και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τα ποσοτικά για να εγγυηθούμε τον ε, διαπολιτισμικό πλουραλισμό. Νομίζω και ότι ο κύριος Χαουρέγου ζήτησε το λόγο. Ναι. Απλώς για να πω ποια είναι η θέση της ομάδας μας σε σχέση με τις ε, θέσεις που εκφράζει ο συγητής. Συμφωνούμε απόλυτα με τις διάφορες τοποθετήσεις και με τις διάφορες τροπολογίες που κατέθεσε ο Πέθυνος επί του προπολογισμού, αλλά είμαστε κατά της, ε, των ε, επιχειρημάτων που αναφέρονται για να διαγραφούν κάποια κονδύλια που δίδονται στον προϋπολογισμό και έχουν σχέση με την επικοινωνία προς τους πολίτες για το τι ακριβώς είναι η Ευρώπη. Και πολλές φορές πρέπει να πω ότι υπάρχει κάτι το παράλογο σε αυτά τα οποία ζητούν κάποιοι συνάδελφοι που έχουν καταθέσει τροπολογίες. Έχουμε το κείμενο, έχουμε το σχέδιο γνωμοδότησης στο δεν, το οποίο συντάχθηκε πριν να κατατεθούν οι τροπολογίες. Στην τροπολογία των κυρίων Καμάλη και Φόξ, όταν γίνεται συζήτηση για ένα κείμενο στην τροπολογία 3, ότι είναι απαραίτητο να φτιάξουμε μια πολιτική επικοινωνίας για να μπορέσουν ε, να συνειδητοποιήσουν ε, οι πολίτες καλύτερα τι σημαίνει η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Μας ε, λένε οι εισηγητές ότι πολλές φορές εκεί αναφέρονται και τα μειονεκτήματα των αναγκασμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τώρα αυτό μου θυμίζει το εξή. Εάν μια χώρα στην πολιτική του, στο σύνταγμά του, προτείνει, υποθετικό είναι, στις ε, διάφορες περιοχές του να χωριστούν και προτείνει μόνο τα, και μιλήσει μόνο για τα πλεονεκτήματα, κάνει κάτι το παράλογο. Σε τέτοιου είδου λοιπόν τροπολογίες πρέπει να πω ότι αναφέρονται στόχοι οι οποίοι πολλές φορές είναι εντελώς αντίθετοι προς τον γενικότερο στόχο της ε, Ενωπής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό τέτοιου είδους τροπολογίες εμείς θα τις απορρίψουμε. Εάν δεν υπάρχουν άλλοι που θέλουν να λάβουν το λόγο, ιδίω η ηγετή εκφράστηκε, μπορούμε να περάσουμε στην ψηφοφορία. Ψηφίζουμε λοιπόν την τροπολογία 6508, το αρθρο 150607 σε σχέση με την Ευρώπη των πολιτών. Λοιπόν, ποιοι είναι υπέρ. Παρακαλώ να σηκώσουν το χέρι. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι απορρίπτεται, δεν νομίζω ότι χρειάζεται επαλήθευση. Άρα η 0667 απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τώρα την επόμενη τροπολογία 6500 επί του ίδιου άρθρου. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την τροπολογία 6507 Ζων Λαμπέρ στο άρθρο 150667 σε σχέση με τον οίκο της Ευρωπαϊκής Κοινωνίας των Πολιτών. Όπως τροποποιήθηκε. Ποιοι τάσσονται υπέρ, δυνατάσεως της χειρός. Έχετε το λόγο. Παρακαλώ, σηκώστε χέρι. Σηκώστε το χέρι. Ποιοι τάσσεστε υπέρ. Να επαληθεύσουμε. Κατά. Εγκρίνεται. Εγκρίνεται. Μία αποχή, μία αποχή, εντάξει. Δύο αποχές. Εντάξει. Πρέπει κάθε φορά να αναφέρω τους αριθμούς, θέλετε, εντάξει. Εντάξει, εντάξει. Υπάρχουν δύο αποχές, λοιπόν. Εντάξει. Α, τρεις, τρεις. Ποιοι απέχουν. Τρεις αποχές. Ευχαριστώ. Εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στην τροπολογία 6.509 σε σχέση με το άρθρο 16.03.01 ε, Messerschmitt υπέρ κατά Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε την τροπολογία 6501 του εισηγητή. Υπέρ. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Ε, ξεχνάω τις αποχές λέει ο πρόεδρος. Το αποτέλεσμα είναι πρόδειλο, επομένω δεν χρειάζεται πάντα. Τέλος πάντων. Θέλετε το λόγο? Μία αποχή. Ωραία. Ωραία. Εγκρίνεται, όπως και να έχει. Ψηφίζουμε την τροπολογία 6510. Μόρτεν Μέσερσμιτ για το επί του άρθρου 160302. Υπέρ, παρακαλώ, διανατάσεως. Κατά. Αποχές. Καμία αποχή. Απορρίπτεται. 6502 του εισηγητή. Επί του ιδίου άρθρου 160302. Υπέρ. Κατά. Τέσσερις αποχές. Απορρίπτεται. Α, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε, λέει ο πρόεδρος, εγκρίνεται, με συγχωρείτε. Τροπολογία 6511. Μόρτεν Μέσσερ Σμιτ, επί του άρθρου 160304. Υπέρ, παρακαλώ. Υπέρ. Βλέπω ότι έχουμε και δύο εκπροσώπους ε, των μη, από τους μη εγγεγραμμένους. Ο αναπληρωτής δεν μπορεί να ψηφίσει, μόνο το πλήρες μέλος. Εν πάση περιπτώσει απορρίπτεται. 6503 ε, λέει ο πρόεδρος, αλλά τον διακόπτει η γραμματεία. Sì, vabbè, allora vogliamo ripetere il voto per chiarezza. Siamo all'emendamento. Βρισκόμαστε στην 65-11, ποιοι τάσσονται υπέρ. Υπέρ, παρακαλώ. Πρόεδρε, νομίζω θα πρέπει να ολοκληρώσουμε την προηγούμενη ψηφοφορία. Uh, Την 6511 δεν την έχουμε ολοκληρώσει. Ε, Μα γι' αυτό, επειδή άκουσα τις ε, παρατηρήσεις σας, είπα ας ψηφίσουμε την 6511 εκ νέου. Γιατί από ό,τι θυμάμαι, δεν είχε ταχθεί κανείς κατά. Λοιπόν, υπέρ της 6511 από την αρχή που αφορά το άρθρο 16.03.04. 65.11. Παρακαλώ, διανατάσεως. Υπέρ, υπέρ. Ποιοι τάσσονται υπέρ. Οι φαβορεύολοι... Υπέρ της 65.11. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 5, 4 sono, 5. 5, eh Κατά. 18. Αποχές. Nessuno astenuto. Κανείς. Απορρίπτεται λοιπόν 65-11. 65-03 του εισηγητή. Πάντα επί του άρθρου 16-03-04. Ποιοι τάσσονται υπέρ. 18 υπέρ κατά πέντε αποχές κανείς, άρα εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στην εξέταση του πρώτου τμήματος που αφορά το Κοινοβούλιο. Α, καταψηφίσατε. Ποιος καταψήφισε που δεν έλαβα υπόψη. Ε, ε, ε, ε, ε, ναι. ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε πρίμα Τμήμα 1. Κοινοβούλιο. Άρθρο 402. Τροπολογία 6512. Μόρτεν Μέσερ Σμιτ. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Κανείς απορρίπτεται. Λοιπόν,

σε σχέση με το άρθρο 403 συνεισφορές στα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα. Γκουαλτιέρη Γκουρμάι, Α, με συγχωρείτε. Μόρτεν Μέσερ Σμιτ, λέει ο πρόεδρος. 65-13. Υπέρ. Υπέρ, παρακαλώ. Η γνωστή 5. Κατά. ασθενούτη. Αποχές. Απορρίπτεται. Οι απέχοντες βρίσκονται σε προνομιακή θέση, λέει ο πρόεδρος. Βρισκόμαστε στο άρθρο 403 του τμήματος 1, τροπολογία 6506. Συνσφορές σε Ευρωπαϊκά Πολιτικά Ιδρύματα. Υπέρ παρακαλώ.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 Τώρα εξετάζουμε τις τροπολογίες στη γραμμοδότηση. Να, να δώσουμε ένα έπαθλο στον ε, κύριο Μέσσερ Σμιτ, διότι δεν εγκρίθηκε τίποτα από τα δικά του. Εν πάση περιπτώσει, θα δώσει μάχη μέχρι τέλους, όπως και να έχει γιατί πολλές φορές ε, δεν αξίζει μόνο η νίκη, αλλά και όλη η συλλογιστική που αναπτύσσουμε για να πείσουμε την πλειοψηφία. Τώρα έχουμε οκτώ τροπολογίες στην ε, παράγραφος, παραγράφους, λοιπόν παράγραφος 1, τροπολογία 3, Καμάλ Φόξ, υπέρ. Ε, Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 2. Τροπολογία 4. Αν μπλοκ. Αν συμφωνείτε, αν συμφωνείτε μόνο, λέει ο πρόεδρος. Δεχόσαστε ψηφοφορία αν μπλοκ. Um, Μπορούμε μέχρι την 7 αν μπλοκ. 7. Ευχαριστώ. Συμφωνείτε όλοι. Ψηφίσαμε την 3 της παραγράφου 1. Τώρα ψηφίζουμε τις 4, 5, 6 και 7. Παράγραφοι 2, 3, 4 και 5. Μέχρι την 7. Ε, abbiamo chiesto, abbiamo detto di votarlo separatamente. Mm. C'è una richiesta di voto separato, così? Ah. Όχι. Είπα ότι θέλω χωριστή ψηφορία στην 8. Άρα 4 με 7 on block. Αυτό είπαμε πρόεδρε. Εντάξει, εντάξει, με συγχωρείτε, εγώ κατάλαβα λάθο. Eh? Άρα περιλαμβάνουμε και την 7. Ωραία, εγώ δεν είχα καταλάβει καλά, λέει ο πρόεδρο. Ποιοι είναι υπέρ αυτών των τροπολογιών, on block. Και contrario. Κατά είναι Αποχές. Άρα ή απορρίπτονται, λέει ο πρόεδρος. Άρα τώρα ψηφίζουμε την 8 της Μαριέτας Γιαννάκου επί της παραγράφου 5α. Κολέγα Σέφλιν. Σέφλιν. Θα ήθελα να πω ότι είναι προφορική τροπολογία, επί της οποίας συμφωνήσαμε νωρίτερα, σε σχέση με την ευημερία ως προς την ελευθερία, αυτή την αντικατάσταση. Ναι, ναι, το θυμάμαι κι εγώ. Ψηφίζουμε την 8, την προφορική. Ποιοι είναι υπέρ. και κοντράριο. 14 υπέρ, κατά. 8 κοντράριο. Και συστήνε. Αποχές. C'è un voto finale. Έχουμε και την τελική ψηφοφορία επί αυτού του σχεδίου νομοδότης όπως έχει τροποποιηθεί. Ποιοι είναι υπέρ. 18. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται λοιπόν. 18 έναντι 5. Άρα κλείνουμε και να συγχαρούμε τον κύριο Σέπφλιν. Τελειώσαμε λοιπόν με τα σημεία 9 και 10. Ecco, 11. Βρισκόμαστε στο 11, μάλλον στην, α, στο χρονοδιάγραμμα το οποίο έχει διανεμηθεί το χρονοδιάγραμμά μας. Οι εκπρόσωποι των ομάδων δέχτηκαν τις προτάσεις της Προεδρίας. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, έτσι ορίζεται. Άρα όσοι θέλουν να πάνε να καπνίσουν εκτός αιθούσης μπορούν. Τελευταίο σημείο. Η ημερομηνία της προσεχής συνεδρίασης. Βρυξέλλες βεβαίως. 6 Οκτωβρίου, 9 με 12.30, 3 με 6.30. Συμφωνείτε? Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, έτσι ορίζεται. Σας ευχαριστώ πολύ και γεια σας.